Okay. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση. Θα συνεχίσω στα Σουηδικά. Hej uh, Καλώς ήρθατε και πάλι λοιπόν στην συνεδρίασή μας. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε πρώτα την έγκριση της ημερήσιας διάταξης και τα αιτήματα τροποποίησης που έχουν τεθεί. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη ως έχει. Ανακοινώσεις Προέδρου το δεύτερο. Θα μπορούσα να σας αναφέρω σχετικά τα εξής. Πολλοί στην δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχουν εκφράσει μεγάλο ενδιαφέρον σε όλα όσα συσχετίζονται με την εκστρατεία One Billion Rising. Ένα δίσα ε, και αυξανόμενο επιπλέον και υπάρχει ενδιαφέρον για όλες τις εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες και στο μεσημέρι 12 η ώρα θα έχουμε μια εκδήλωση στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν οι ευρωβουλευτές και είναι κάτι πολύ καλό να συμμετάσχει κανείς σε αυτή την εκδήλωση διότι υπάρχει η συνδιοργάνωση από πλευρά της κυβέρνησης. Η κυρία Πάκα λάβει τον λόγο, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού. Αποφασίσαμε όμως να έρθει πριν από την ψηφοφορία, πριν από τις ψηφοφορίες, τότε θα έρθει και δεν θα λάβει τώρα φυσικά τον λόγο και θα μας ανακοινώσει κάποια πράγματα. Τρίτον, μπορώ να σας αναφέρω ότι ο χώρος για αύριο, για την δημόσια ακρόαση από κοινού με την άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή άλλαξε. Είναι 4Q2 Εκεί θα διεξαχθεί η ακρόαση 4Q2 στο κτίριο Άνταλ Ιωζεφ Και περνάμε στο σημείο 3 της ημερησίας διάταξης που είναι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα ΆΙΓΕ μεταξύ ανδρών και γυναικών και ως ήθιστε συνεργαστήκαμε στενά με το Ίδρυμα αυτό, το Ινστιτούτο ΆΙΓΕ και πάρα πολλά στοιχεία και πραγματικά γνώση διοχετεύει και παρέχει η, ε, ο θεσμός αυτός, ο οργανισμός αυτός. Έχουμε αποφασίσει και συναντώμεθα σε τακτά χρονικά διαστήματα με την επικεφαλής ε, της ΆΙΓΕ. Η Βιργίνια είναι παρούσα και θα συζητήσουμε για το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και όλα αυτά θα γίνονται πολύ πιο τακτικά και πολύ πιο συχνά από ό,τι κατά το παρελθόν. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαστε εδώ κυρία Βιργίνια Λάγκμπακ. Θα έχετε περίπου 20 λεπτά για την παρέμβασή σας και θα έχουμε χρόνο για τις ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Καλώς ήρθατε και πάλι θερμά, έχετε τον λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και είναι πραγματικά, όπως λέμε κάθε φορά, μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και πραγματικά αδειμονούμε να ακούσουμε τις παρατηρήσεις των Ευρωβουλευτών Δυστυχώς έχω βραχνιάσει και δεν θα μπορέσω να αποδώσω καλύτερα. Αλλά πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω γενικότερα ότι εφέτος από πλευράς μας αυτό το οποίο πραγματικά ολοκληρώνουμε στη δράση μας και μπορούμε να το πούμε αυτό διότι προπαρασκευάζουμε την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και σε σχέση με αυτό που έγινε και σε σχέση με πέρσι είναι ότι ξεκινήσαμε μια επισκόπηση των υπολοιπόμενων δραστηριοτήτων σε σχέση με τα όσα σχεδιάζαμε για τον κανονισμό στα κυριότερα έγγραφά μας, δηλαδή σε σχέση με, τον, το παράρτημα και τα στοιχεία για τους ποιοτικού δείκτες και σε σχέση και με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ισότητα και θα έχετε ακούσει ότι συζητούμε και χρησιμοποιούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό τον ίντεξ, αυτό τον κατάλογο και σε σχέση με το κέντρο μας και το δίκτυο που έχουμε δημιουργήσει. Εξακολουθούμε να αναζητούμε τις καλύτερες δυνατότητες και διάβλους για εφέτος αυτό που θα κάνουμε είναι θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε και να δούμε πόσο αποτελεσματικά είναι όλα αυτά. Ποια είναι η χρήση ε, στα όσα εισάγουμε για ένα σύστημα υποπτίας και παρατήρησης. Πόσοι χρήστες ε, για αυτούς τους πόρους ε, υπάρχουν. Υπάρχουν αρκετοί ευρωβουλευτές που και σε σχέση με πληροφορίες που ζήτησαν έγινε η προσπάθεια να υποστηριχθούν Θέλουμε να δούμε σε, ποια, σε ποιο εύρος θα πρέπει να γίνονται όλα αυτά. Εξαρτώνται από την εποπτεία εφέτος ποια είναι η χρήση και ποια είναι η εμβέλεια αυτής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του ε, συστήματος τεκμηρίωσης. Την προσοχή σας θα ήθελα να επιστήσω και στις διαφάνειες. Ακόμα και αν δεν αφορά την φετινή χρονιά, είμαι υπερήφανη και αυτό θα είναι τμήμα και της έκθεσής μας για πέρυσι βέβαια, αλλά όπως βλέπετε, ξεκινώντας από τον Ιούνιο ήδη του 2010, πώς χρησιμοποιήθηκαν τα κονδύλια μας σε σχέση με την αρνητική εξέλιξη των πραγμάτων η υλοποίηση των δράσεων προχώρησε με πολύ θετικό τρόπο και καθότι μπορείτε να δείτε για εφέτος και για πέρυσι μπορέσαμε πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε και να εκτελέσουμε τα κονδύλια του προϋπολογισμού στα επίπεδα που είχαν προσχεδιαστεί. Έχουμε το δυναμικό και την ικανότητα λοιπόν μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων σε σχέση με τα όσα είχαμε κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους έχουν μειωθεί αυτά τα κονδύλια τώρα βέβαια αλλά αν δει κανείς ευθύς εξ αρχής ξεκινώ με αυτό διότι έχω πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μου. Αυτό που βλέπουμε και πραγματικά αυτό που ε, χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό και το βλέπουμε αυτό. Η πρόσθετη αξία είναι πάρα πολύ μεγάλη σε υψηλό επίπεδο για τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων όχι μόνο για το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και στα κράτη-μέλη υπάρχει εμπλοκή και η Επιτροπή συμμετέχει. Είναι οι εκθέσεις που υποβάλλουμε στις Προεδρίες. Εφέτος ολοκληρώνουμε δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, γι' αυτό δεν θα καταδείξω κάποια στοιχεία, αλλά βρισκόμαστε σε μια φάση πολύ ε, με πολύ ενδιαφέρον για τις δραστηριότητές μας, για την ελληνική προεδρία, γυναίκες και οικονομία. Προετοιμάζουμε τρεις ε, συνολικά δείκτες, ε, τρεις δείκτες και εννέα κεφάλαια, εννέα τομείς, θα υπάρξει η ε, πλήρης έκθεση, αλλά ένα από τα προσωρινά συμπεράσματα είναι ότι αναλύουμε την ε, αντιστοιχεία σε σχέση με την πλήρη απασχόληση στην αγορά εργασίας και σε σχέση και με την ε, ομάδα υψηλών αξιωματούχων για την ισότητα των φύλων στην Αθήνα, αν μετρήσει κανείς τους στόχους ε, της Λισαβόνας ε, για την απασχόληση 75% επίτευξη απασχολησιμότητας και αν δει κανείς την εικόνα και αν δει κανείς την αντιστήχηση με τα μέτρα που λαμβάνονται σήμερα, τότε η κατάσταση δεν είναι καλή και είναι ακόμα αρνητικότερη για τις γυναίκες. Και αυτό που καταδεικνύεται και είναι για τους υπεύθυνου για την λήψη αποφάσεων, το σημαντικό είναι πού μπορεί να υπάρξουν και να δημιουργηθούν τέτοια μέτρα για να προαχθεί αυτός ο τομέα και θα μπορούσε αυτό να είναι χρήσιμο και για τα διάφορα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κάτι άλλο που αναλύουμε είναι δείκτε για το επιχειρήν, για την επιχειρηματικότητα για τι γυναίκε και για την απασχόληση. Και ε, βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει ένα τομέα που πολλά πρέπει να γίνουν και στι μικρομεσαίες επιχειρήσει και σε σχέση με το επιχειρήν, την επιχειρηματικότητα. Στι χώρε εκείνε όπου η αυτοαπασχόληση είναι ιδιαίτερα υψηλή για τι γυναίκε, δείχνουν τα πράγματα ότι η κατάσταση κατάσταση είναι πολύ αρνητική για τις γυναίκες και όπως αναφέρθηκε στην έκθεση είναι μια παγίδα που δημιουργείται για τις γυναίκες και αυτοπαγιδεύονται εκεί. Είναι δύσκολο λοιπόν να αποκληθεί κάτι τέτοιο επιχειρηματικότητα. Αυτή η έκθεση λοιπόν σε πολύ θετική χρονική συγκυρία υποβάλλεται και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Και σε το ε, εθνικό επίπεδο θα συζητηθούν τα θέματα αυτά και ελπίζω ότι και η Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γυναικών του Ευρωκοινοβουλίου θα μπορέσει να δει και να εξετάσει πώς θα ερμηνεύονται και θα ερμηνευτούν αυτά τα στοιχεία σε σχέση με τα κράτη-μέλη, σε σχέση με την ε, δική μας έκθεση. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Ιταλική Προεδρία. Μια πρώτη αναθεώρηση. Τι επετεύχθη κατά τις ε, δύο πρώτες δεκαετίες από πλευράς των ε, κρατών μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την πλατφόρμα των Ηνωμένων Εθνών για την δράση υπέρ της ισότητας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα συλλέξουμε τα στοιχεία αυτά δεν θα, υπάρχει ε, κάποια διαφορετική παρουσίαση. Θα ακολουθήσουμε και το πρότυπο το σουηδικό του 2009. Θα προσθέσουμε κάποιες θετικές ε, πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί οι βέλτιστες πρακτικές είναι κάτι το οποίο ζητείται όλο και συχνότερα από τους εμπλεκόμενους και τα κράτη-μέλη για να εξεταστεί και να δούμε πώς μια χώρα είχε τις α ή β επιδόσεις και σε τι οφείλονται αυτές οι επιδόσεις. Θα υποβληθούν αυτά στην έκθεση ύστερότερα, θα είναι όμως ένα πολύ σημαντικό τμήμα του έργου μας. Εδώ βλέπετε μία διαφάνεια, απλά για να ε, υπενθυμίσω ότι πέρυσι και ο κύριος Γκούσταυσον ε, ήταν παρόν, όταν ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία Index για τον κατάλογο αυτό πέρυσι, για το τι θα κάνουμε τώρα εφέτος. Αυτό που έχουμε είναι ότι βρισκόμαστε ήδη σε μια εβδομάδα ξεκινά το έργο με τις συζητήσεις ε, πραγματογνωμόνων και ειδικών για την βία, αντιμετώπιση της ε, ε, βίας. Ε, δεν υπήρχαν κάποια στοιχεία σε σχέση με αυτά τα θέματα. Είναι ειδικά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ζητήθηκε να δοθούν συμβουλές πώς θα μπορούσαν να διευρυνθούν αυτά τα ζητήματα, σε ποιους τομείς θα μπορούσαν με τους κατάλληλους δείκτες να μετρηθούν τα θέματα αυτά. Έχουμε συζητήσει το θέμα πώς μπορούν να προσθεθούν οι δείκτες για την επικέντρωση στην εργασία και τη βία και σε σχέση με ε, ποιοτικά επίπεδα που μπορούν να επιτευχθούν με αυτούς τους δείκτες συζητώντας για τα θέματα ηλικίας για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι για τους ε, ε, πρεσβύτες, τους νεότερους, ε, τους μετανάστες θα μπορέσουμε να δούμε πώς ανανεωμένοι δείκτες, νέοι δείκτες μπορούν να εμπλουτίσουν τον κατάλογο και το, την φαρέτρα μέσων που έχουμε και σε σχέση και με τους παρόχους των στοιχείων αυτών και σε σχέση με συνεργασία ε, συνεχίζεται και το έργο από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη βία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αλλά και διάφορα κράτη-μέλη και οργανώσεις θα εμπλακούν και θα συμμετάσχουν. Αυτό που εστιαζόμαστε φέτος να κάνουμε είναι να δημιουργηθούν αξιόπιστοι ε, δείκτες και να μπορέσει αυτό το εγχείρημα να προχωρήσει και την επόμενη χρόνια του χρόνου ένας τομέας όπου πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ε, θετική συλλογή πόρων και στοιχείων για να αναλυθούν αυτά τα στοιχεία θα είναι η ε, δειγματοληπτική προσπάθεια για τα στοιχεία για την ε, βία αναφύλω και θα έχουμε και πρόσβαση σε μικρο στοιχεία, micro data, και θα μπορέσουμε να αναλύσουμε ποιοι δείκτες θα μπορέσουν να εκπονηθούν και για τον κατάλογο index αλλά ε, και για το έργο μας ε, για την ε, εξειδικευμένη μορφή βίας σε σχέση με τις γυναίκες σε σχέση με το φύλλο. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε λοιπόν σε αυτές τις παραμέτρους και ολοκληρώνοντας μπορώ να πω ότι έχουμε διάφορες μελέτες που υποβάλλονται και ολοκληρώνονται. Φέτος ολοκληρώνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για τις διοικητικές πηγές ως στοιχεία θα είναι χρήσιμο αυτό το εγχείρημα για οποιουσδήποτε εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε ποια επίσημα στοιχεία υφίστανται σε σχέση με τη βία ώστε όλοι να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για το έργο τους ε, ξεχωριστά και να δούμε τι μπορεί να γίνει και σε σχέση με τη χρήση με τους δείκτες. Και φέτος θα ολοκληρώσουμε μια σχετικά μικρή μελέτη αλλά ενδιαφέρουσα παρόλα αυτά για το κόστος της βίας το κόστος της βίας όπως γνωρίζετε είναι πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα να μετρηθεί, να σταθμιστεί. Θα δούμε ποιες προσεγγίσεις μπορούν να ακολουθηθούν για την καταμέτρηση, την ε, αξιολόγηση του κόστους της βίας και για να, την αναζήτηση προτάσεων και συστάσεων ποιες μέθοδοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν ή αναλύθηκαν σε σχέση με την καλύτερη αποτελεσματικότητά του όσον αφορά το κόστος σε σχέση με το όφελος για να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη-μέλη. Θα ακολουθήσει και μία μελέτη για τον, για τον ακροτηριασμό ε, των γενετικών οργάνων γενετήσιο ακροτηριασμού και αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα παρέμβασης μετά από την μελέτη που συντάχθηκε για τους ακροτηριασμούς αυτούς που υφίστανται ε, γυναίκες. Και ολοκληρώνοντας σε σχέση με τα θέματα βίας, θέλω να πω ότι θα αναλύσουμε όλα τα στοιχεία φέτος, όλα όσα είναι διαθέσιμα και υφίστανται και για την δειγματοληπτική μας αυτή δράση, την μελέτη μας και θα προετοιμάσουμε προτάσεις και σχέδια για το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εγκριθούν κατά τα τέλη του έτους, πώς δηλαδή μακροπρόθεσμα μπορεί να θεμελιώνεται και να διαμορφώνεται η καταπολέμηση της βίασης βάρος των γυναικών. Είναι ένα θέμα το οποίο πολλές φορές το αποφεύγουν ε, οι ε, άνθρωποι γιατί είναι πολύ δύσκολο και να το προσεγγίσουν και για να γίνει απόλυτα κατανοητό. Αυτό που σχεδιάζουμε είναι μια αμφίδρομη δράση ηλεκτρονικά στο δίκτυο ένα εργαλείο ή μέσο ώστε να υπάρχει το θέμα της ε, ισότητας των φύλων πιο ολοκληρωμένα μέσα σε αυτό. Δεν μπορούμε πιο εξειδικευμένα να αναπτύξουμε την πιο δημοφιλή προσέγγιση πρόσβασης και κατανόησης άμεσα. Αυτό θα είναι πιο εξειδικευμένο, απαιτεί περισσότερο χρόνο. Θα γίνει αυτό όμως ένα πρώτο βήμα σε μια πρώτη φάση και μετά θα ακολουθήσει η πρωτοβουλία αυτή που θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη για τις επιπτώσεις της ισότητας μεταξύ των ανδρών και γυναικών. Η ισότητα των δύο φύλων είναι υποχρέωση που έχουν επομιστεί τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτού σχεδιάζεται πολιτική και λαμβάνονται ε, από τους αρμόδιους οι αντίστοιχε αποφάσεις. Θα είναι λοιπόν μια, ας το πω έτσι, συνεισφορά στι στις βέλτιστες πρακτικές και θα είναι διαθέσιμα όλα αυτά και τομεακά. Διότι θέλουμε να επισέλθουμε τομεακά, εξειδικευμένα στους διάφορους τομείς. Θα είναι πιο εύκολο και να γίνεται κατανοητό αυτό για τους πολίτες τομεακά. Διάφορες πληροφορίες για τις διάφορες και διαφορετικές πολιτικές για να αποκτήσουν μια πρόγευση, μια πρώτη εντύπωση περί τίνος πρόκειται. Και θα ξεκινήσουμε και μια τέτοια προσέγγιση για ε, φέτος ήδη και συμφωνήσαμε στο Συμβούλιο μας να υπάρξει μια σε βάθος μελέτη τι γίνεται σε σχέση με την έρευνα και καινοτομία για παράδειγμα, σε σχέση με την ισότητα. Είναι ένας ευρύτατος τομής, θα συναντηθούμε με αρμόδια θεσμικά όργανα να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τα θέματα της ισότητας όσον αφορά την καινοτομία για παράδειγμα. Ποιες αλλαγές θα συνεπαγόταν κάτι τέτοιο. Αυτό είναι, αυτά είναι τα σχέδιά μας μέχρι τώρα. Και για την ισότητα των φύλων είναι πολύ σημαντικό αυτό αυτό ως εγχείρημα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο δραστηριοτήτων ελπίζω ότι θα μπορέσουν να ενταχθούν και να ευδοκιμήσουν αυτά. Αυτό που κάνουμε φέτος και μόλις ξεκινήσαμε είναι αυτό το οποίο επιθυμούμε περισσότερα να εξευρεθεί. Μια προσέγγιση ώστε με οποιονδήποτε συναντάτε κανείς, ο οποίος μπορεί να μην είναι ο πιο άμεσα ενδιαφερόμενος για τα θέματα ισότητας, να μπορούμε να συνεισφέρουμε αποδεικνύοντας, καταδεικνύοντας ότι ορίστε είναι σημαντικό να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων και έχουμε δεσμεύσει και έχουμε και έξι ε, έρευνες που έχουν συνταχθεί θα αναλυθούν και θα αναλύσουμε τα στοιχεία και τα τεκμήρια προτού καταλήξουμε σε πιο εξειδικευμένες προτάσεις και σε σχέση με τις υποένταξη χώρες ε, υπάρχει και ε, σε αυτές πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ισότητα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με αυτές τις πρωτοβουλίες και ε, μελλοντικά και προσεχώς. Θα, αυτά τα οποία ανέφερα για τους πόρους στην αρχικά Υπάρχουν ε, πόροι και δυνατότητες ε, για στρατός και σε συνεργασία με τις ε, βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφόρησης και ενημέρωσης και από πλευράς Κοινοβουλίου έχουμε διάφορες υπηρεσίες που συνεργάζονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο ενός σε εισαγωγικά τεκμηριωμένου θησαυρού μιας ολοκληρωμένης φαρέτρας πανοπλίας στοιχείων ώστε να μπορέσουν τα στοιχεία για την ισότητα να διαχέονται περισσότερο. Και κάνοντας λόγο και για τους άνδρες, ένα μικρό ποσοστό, 10% συνολικά σε σχέση με τις δραστηριότητες, όμως η προσπάθεια προσέγγισης σε σχέση με τους άνδρες για τα θέματα ισότητας είναι κάτι περισσότερο ε, που αφορά την δημιουργία εταιρικών σχέσεων με ε, ε, εκπροσώπους του πληθυσμού άνδρες που έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα άσκησης επιρροής ε, επ' αυτόν. Έχουμε προσκαλέσει διάφορους σημαντικούς ε, πολιτικούς άνδρες ώστε να προσθέσουν τις προσπάθειές τους ως πρωτοβουλίες στην ευρύτερη εκστρατεία κατά της βίας εις βάρος των γυναικών. Και με πολιτικούς υπουργούς αυτά είναι αυτά τα οποία σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή και είναι στη διάθεσή μας σε σχέση με σημαντικά συμμετέχονται συμμετέχοντες ε, εξέχουσες προσωπικότητες που μπορούν να ασκήσουν την επιρροή τους και να επηρεάσουν τις εξελίξεις. Αυτό εκπονούμε σε μια πρώτη προσέγγιση, σε μια πρώτη φάση. Ιστερότερα θα δούμε πώς μετεξελίσσεται αυτό. Η κυριότερη προσέγγιση είναι η καταπολέμηση της βίας. Εκεί θέλουμε να επικεντρωθούμε, ξεκινώντας αυτή τη συνεργασία μας σε μια εταιρική σχέση με τους άντρες. Αυτά κατά το μάλλον οι ήτων είναι με τα παλαιότερα και νεότερα στοιχεία, τα στοιχεία εκείνα τα οποία διαμορφώνουν το έργο μας. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας, κυρία Λάγκμπακ. Ε, και να ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση. Θα ξεκινήσουμε με τις δικές μου ερωτήσεις. Καταρχάς, να κρατήσουμε ως πολύ σημαντικό ποσοστό το 55% μιλήσατε για τη δυσκολία υπολογισμού. Τη δυσκολία του να υπολογίσει κανείς. Όμως, εάν σκεφτείτε πόσο δύσκολα γίνονται αυτοί οι υπολογισμοί, πόσο δύσκολα καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε αυτά τα ποσοστά, φαντάζομαι ότι τα ποσοστά είναι ακόμη χαμηλότερα εφόσον μιλάμε για τη μερική απασχόληση. Και αν ληφθεί και αυτή, και αυτή η υπόψη. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο κανείς να συνδυάσει αυτά τα στοιχεία εάν σκεφτούμε ότι διαφορετικές σταδιοδρομίες μπορεί να ακολουθήσει μια γυναίκα. Από το να είναι διευθύντρια κάπου μέχρι το να ακολουθήσει μια πολιτική καριέρα. Στην ε, διατύπωση λοιπόν αυτή του Συμβουλίου δεν είναι σαφή τα πράγματα. Εδώ λοιπόν θα έπρεπε να ε, εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και να σας πω ότι ο δείκτης για την ισότητα είναι ένας δείκτης πολύ σημαντικός. Τον βρίσκω ένα εξαιρετικό εργαλείο. Και εγώ τον έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές στο παρελθόν για να κατανοήσω καλύτερα το πώς έχουν τα πράγματα. όχι μόνο σε επίπεδο κρατών μελών, σε εθνικό επίπεδο, αλλά για να καταλάβω και πώς εξελίσσεται η ισότητα των φύλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σίγουρα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι εξελίξεις τις οποίες αναφέρατε και ελπίζω ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε όντως να καλύψουμε και τη συνιστόσα της βίας κατά των γυναικών. Τώρα να περάσουμε στους συναδέλφους και στις συναδέλφους. η έρευνα που θα κάνετε για τη βία αναφύλλω ή ως προς το φύλλο. Θα πρέπει να σκεφτούμε και το κόστος της. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Εγώ θα μπορώ να ε, αξιοποιήσω όμως τα δεδομένα που θα συγκεντρώσετε από την ε, πολιτική σκοπιά ή μόνο οι ερευνητές ε, θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να είναι και για μας εύληπτα. Αλλά επίσης θα θέλαμε να καταλάβουμε και πόσο θα κοστίσει μια τέτοια έρευνα. Και μια ακόμη ερώτηση. Αυτά τα εργαλεία τα οποία αναφέρατε για το mainstreaming, για την ε, συμπερίληψη αυτών των δικτών είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να, να συμπεριλαμβάνονται στο πολιτικό σύστημα. Όπως είπατε πρέπει να δούμε αυτά τα επιμέρους θέματα. διότι φαίνεται κάποιες φορές ότι είναι δύσκολο να καλύψουμε και την διάσταση της ισότητας των φύλων, όμως Εκ των υστέρων βλέπουμε ότι στην πράξη ισχύει ίσω το αντίθετο. Γι' αυτό πρέπει τα διδάγματα που διαθέτουμε να ξέρουμε να τα αξιοποιούμε. Ελπίζω λοιπόν ότι όταν θα μας ε, παρουσιάσετε τέτοιου είδους νέα εργαλεία και εμείς από την πολιτική σκοπιά θα μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε στο πολιτικό μας έργο. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτές ήταν οι δικές μου ερωτήσεις και να ξεκινήσουμε την συζήτηση με την κυρία Γκάμπριελ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Λάνμπακ, ευχαριστούμε για την προσέλευσή σας σήμερα. Ευχαριστούμε και για αυτή τη λεπτομερή παρουσίαση. Καταρχάς, να κάνω κάποιες επισημάνσεις επί της Παρουσία πρώτα απ' όλα και μετά επί της ουσίας. Πρώτα απ' όλα, επί της παρουσίας να σας ε, συγχαρώ για την ε, επίκαιρη δράση σας και γιατί πραγματικά είσαστε ε, γέρο εδώ όταν σας χρειαζόμαστε. Ενημερωνόμαστε διαρκώς για το πώς προχωρούν οι εργασίες σας και σήμερα έχουμε ένα μήνυμα ενθαρρυντικό για το ότι μπορεί να λάβει συστηματικό χαρακτήρα η επικοινωνία μας. Μια επικοινωνία που είναι καλή και πάντοτε σταθερή όταν ετοιμάζει έκθεση ετοιμάζει ετοιμάζει έκθεση Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Γυναικών και οργανώνουμε δημόσιες ακροάσεις. Ε, μια πρώτη ερώτηση για το Ινστιτούτο στη δημόσια ε, κρόαση για την ε, ισορροπία του επαγγελματικού βίου και την ισότητα των φύλων θα, θα είστε κι εσείς εκεί. Διότι στην έκθεση που θα ετοιμαστεί καλό θα είναι να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα αριθμητικά στοιχεία και τα δεδομένα που διαθέτει το Ινστιτούτο παρά ε, μία αξιόπιστα ή μία επαληθεύσιμα στοιχεία. Τώρα επί της ουσίας ήθελα να παρατηρήσω ότι οι μελέτες που προβλέπονται στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας δίνουν έμφαση στην μερική την επιχειρηματικότητα των γυναικών, πρακτικές, τη χρηματοδότηση. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και για μας είναι πολύ χρήσιμα. Είναι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα για να μπορέσουμε όντω να πετύχουμε καλύτερη ισορροπία στην προσέγγιση που έχουμε και εμεί στο δικό μα έργο ω ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή και την προώθηση τη ισότητα των γυναικών. Το ερώτημά μου αφορά τον αντίκτυπο που θα έχει το Eurogender Network, το δίκτυο δηλαδή για την ισότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ποιοι είναι οι στόχοι ακριβώς αυτού του δικτύου και πώς ε, προβλέπετε να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί. Αυτή είναι η βασική μου ερώτηση και πραγματικά να σας συγχαρώ για την δημιουργία του δίκτυ για την ισότητα των φύλων, το Gender Equality Index, ε, είναι μια από τις πιο καλές ε, κινήσεις που έχουν γίνει πρόσφατα και επίσης πολύ καλό το να συγκεντρώνονται στοιχεία για την βία κατά των γυναικών. Και πάλι συγχαρητήρια για την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων με τους άντρες, τι καλέ σχέσεις που αναπτύσσονται με τους άντρες, γιατί εκείνοι θα γίνουν οι μεγαλύτεροι υπερασπιστέ των δικαιωμάτων των γυναικών και αυτό το διαπιστώνουμε και στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπιλμπάου, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και για την παρουσίαση, την ενημέρωση. Έχω διάφορες ερωτήσεις. Η γενική εκτίμηση νομίζω ότι είναι απολογισμός έντονης δραστηριότητας από το Ινστιτούτο σας. Ξέρω και τις δυσχέρειες που έχετε και θέλω να εκφράσω τη στήριξη και τα συγχαρητήριά μου. Για την έκθεση στην οποία βρεθήκατε οι γυναίκες και η οικονομία, διαπιστώνω ότι κάθε φορά που εκπονούμε τέτοιες εκθέσεις, το κάνουμε από, με αρνητική προσέγγιση. Δεν λέω ότι πρέπει να παραχαράξουμε τα στοιχεία. Τα στοιχεία για την μερική απασχόληση και πλήρη απασχόληση των γυναικών τα έχουμε αναλύσει επανειλημμένα. Και είναι σαφής η ανισότητα. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, εάν δεν θα έπρεπε να δείτε και με θετικό τρόπο τα θέματα αυτά. Δηλαδή, τα στοιχεία που έχουμε για τα συμβόλαια Αμερικής και πλήρους απασχόλησης σαφώς καταδεικνύουν ανισότητα παντού. Αλλά γιατί να μην ε, τα δούμε και από, τα εξής, ε, από την εξής θετική γωνία. Έχουμε όλο και περισσότερες εκθέσεις που διαπιστώνουν ότι οι γυναίκες ε, στον επιχειρηματικό κόσμο δίνουν περισσότερη καινοτομία, δημιουργικότητα, ε, και μένουν περισσότερο στις επιχειρήσεις. Θα ήταν λοιπόν καλό να έχω τη γνώμη σας από αυτόν, γιατί να μην είναι λίγο πιο ισορροπημένες οι εκθέσεις. Αυτά είναι τα αρνητικά στοιχεία, αλλά για αυτά τα θέματα θα άξε τον κόπο τα κράτη να εμπλακούν περισσότερο στην εργασία, στις συνθήκες εργασίας των γυναικών. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Γιατί να μην μπει και αυτό με στην έκθεση. Δεύτερη ερώτηση. Στην έκθεση που είπατε ότι θα εκπονήσετε με την Τελική Προεδρία τι έχουν κάνει τα κράτα τελευταία 20 χρόνια, θα ήθελα να μου πείτε αν θα περάσετε και σε περιφερειακό επίπεδο. Γιατί εγώ είμαι από τη χώρα των Βάσκων, ξέρετε. Στη χώρα των Βάσκων το 2005 είχαμε ως πρόεδρο έναν άνδρα που είχε ως βασική αποστολή να εγκριθεί ένας νόμος για την ισότητα των φίλων. Και εγκρίθηκε αυτός ο νόμος ε, που ήταν πρωτοπόρος για ε, την ισότητα των ε, φίλων. Από το 1988 έχουμε ένα του που λέγεται Μακούντε και έχει επιτύχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Γιατί λοιπόν να χαθούν τα διδάγματα, η πείρα από τέτοια Ινστιτούτα που μπορεί να λειτουργούν ήδη στις χώρες μας και που δεν είναι εθνικά κρατικά Ινστιτούτα. Γι' αυτό ρωτάω μέχρι σε ποιο επίπεδο θα πάτε. Τώρα για τη συλλογή στοιχείων για την ε, βία με βάση το φύλλο. Υπάρχουν κράτη μέλη της Ένωσης που θεωρούν ότι αυτά τα θέματα είναι ιδιωτικής φύσης και δεν υπάρχουν κανόνες για αυτή. Πρόκειται να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό. Και τι μεθοδολογία έχετε για την ε, συλλογή και αποτίμηση των στοιχείων. Τι στοιχεία θα ζητήσετε. Και τέλος, τέλος. Για τους άνδρες. Είπατε ότι πρέπει να κάνουμε εκστρατεία κατά της βίας. Δεν συμφωνώ και τόσο πολύ με το σύνθημα. Διότι σε τελευταία ανάλυση η βία είναι απόρρια της ανισότητας. Πιο θετικό πιστεύω θα ήταν ε, η καμπάνια μας να είναι υπέρ της ισότητας των φίλων. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα βλέπαμε με γενικότερο τρόπο. Νομίζω ε, το θέμα αυτό. Και έχουμε ήδη θετικές εμπειρίες. Γιατί έχουμε συμφωνήσει ε, στη χώρα των Βάσκων σε μια τέτοια διακήρυξη καλέσαμε και τους άντρες να την υπογράψουν και προέκυψε ε, μια ολόκληρη κίνηση και από πλευρά των ανδρών για την ισότητα των φύλων. Υπήρξε ευρεία συμμετοχή. Γιατί πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι μία από τις ε, θλιβερές επιπτώσεις της ανισότητας είναι η βία κατά των γυναικών. Και πιστεύω ότι τώρα, στον 21ο αιώνα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις νέες αρενοπότητες, όπως λέγονται. Υπάρχουν λοιπόν ε, νέου τύπου αντιλήψεις που οδηγούν σε τέτοιες εκδηλώσεις βίας. Έτσι πιστεύω θα μπορούσαμε να επιτύχουμε περισσότερα σε αυτές τις εκστρατείες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μήπως μπορείτε παρακαλώ να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις σας. Ξεκινώ με τις ερωτήσεις του Προέδρου για το κόστος σε σχέση με τη βία και ποιοι εποφελούνται και ποιοι, ποιες είναι οι ομάδες στόχοι. Η μελέτη αυτή σε μια μικρότερη κλίμακα με σύγχρονες μεθόδους θα χαρτογραφήσουμε πώς σήμερα στα ταυτοποιημένα εντοπισμένα εκείνα πρότυπα και μεθόδους υπολογίζεται με ποιο τρόπο το κόστος και πώς για να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να παρουσιάσουμε στα κράτη-μέλη και στους ε, όσους υλοποιούν αυτές τις πολιτικές τις δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή τους. Αυτό θα είναι η δουλειά των κρατών μελών, των κυβερνήσεών τους. Αν θα θέλει κάποιο κράτος μέλος, μια κυβέρνηση να υπάρξει με βάση αυτά τα στοιχεία να προσθεθούν κονδύλια σε σχέση με τη δράση για τα πολέμηση της βία των γυναικών, αυτό είναι κιόλα και το μήνυμα, στοχεύοντας και στις εθνικές κυβερνήσεις έτσι, αλλά και τα επιχειρήματα, το πώς υπολογίζονται αυτά τα κόστη μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέροντα και για τους ίδιους τους πολιτικούς. Όταν θα υπάρχουν λοιπόν αυτά τα στοιχεία θα υπάρξει μια γενικότερη τοποθέτηση και από πλευρά της Επιτροπής και της Επιτροπής Γυναικών να δούμε πώς ε, προχωρεί αυτό, προχωρά αυτό το πράγμα. Τώρα και για την ισότητα των φύλων ε, πώς μπορεί με ποιο τρόπο και πιο εύκολα να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά. Αυτό που σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή και πάλι είναι περισσότερο για να υποστηριχθούν οι όσοι υλοποιούν επιτόπου στην πρακτική εφαρμογή τους, ε, οι καθημερινά εμπλεκόμενοι, κρατικοί υπάλληλοι, ε, εκείνοι που από πλευράς περιγραφής ε, του έργου τους έχουν και τα θέματα ισότητας στο ευρύτερο έργο τους. Σε σχέση με αυτή τη μελέτη λοιπόν για τους αρμόδιους που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντοπίσουν αυτά τα στοιχεία ε, πιο εύκολα, καθώς και οι πολιτικοί που θα μπορούν να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα πάλι. Είναι μια σε εξέλιξη, υποεξέλιξη, ζωντανή, ενρευστό διαδικασία και θα δούμε τι μπορούμε να προσθέσουμε ώστε να ολοκληρώσουμε βήμα προς βήμα και σε σχέση με τα όσα αναφέρονται από πλευράς ε, Έρικα για την αύξηση του δυναμικού και των δυνατοτήτων ε, για την καταπολέμηση των ανισοτήτων για να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων. Έτσι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε υστερότερα. Αλλά αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε σε εκείνους που πρέπει να επιτελέσουν αυτό το έργο σε αυτή τη φάση. Και για την ερώτηση αν θα, βρεθούμε, θα συμμετάσχουμε στην ακρόαση, δεν γνωρίζω δυστυχώς ποια ακρόαση εννοούσατε στο Ευρωκοινοβούλιο ή ποια ακρόαση. Διότι η ακρόαση που, ε, περί της οποίας πρόκειται αν είναι κάτι το οποίο θα χρειαζόσαστε πληροφορίες και θα χρειαζόσαστε την παρουσία μας, με μεγάλη χαρά να υποστηρίξουμε και εμείς αυτό το εγχείρημα. Αλλά δεν έχω αυτές τις πληροφορίες για κάτι τέτοιο. Αν το χρειάζεστε θα παραστούμε και εμείς με προσώπους μας σε αυτή την ακρόαση. Τώρα, για το Eurogender, το δίκτυο ε, ε, σε σχέση με την Ευρώπη για τα φύλλα για, για ε, εξειδικευμένες δράσεις ε, για τα φύλλα. Τώρα, με συγκεκριμένους πραγματογνώμονες ε, για το gender mainstreaming, την ένταξη του θέματος της ισότητας των φύλων και σε ακροάσεις και όλο και περισσότερο θέλουμε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Γυναικών και άλλοι να διεξα... μπορούν να διεξαγάγουν τέτοιου είδους δραστηριότητες και συζητήσεις πριν από τις ευρωεκλογές. Θέλουμε να υποστηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία ξεχωριστά όπου θα μπορούσαν οι γυναίκες ε, να ε, βρίσκονται στο επίκεντρο, να έχουμε μια καλύτερη αναλογία σε σχέση με την αριθμητική σχέση ανδρών γυναικών σε σχέση με τις γυναίκες. Ένα προς, ε, έχουμε διάφορες συζητήσεις σε σχέση με το Eurogender και που θα εμπλέκουν όχι μόνο εθνικούς ε, πραγματογνώμονες επαΐοντες αλλά και βουλευτές ε, και που θα θέλαμε πάρα πολλοί ευρωβουλευτές από πλευρά των Βρυξελών ε, του Ευρωκοινοβουλίου να συμμετάσχουν και σε σχέση με αυτό το θέμα και τις εκλογές πάλι εξαρτάται και πώς βλέπουμε τα πράγματα αυτά, πώς χρησιμοποιούνται και πώς θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες δράσεις, επικεντρωνόμενοι από αυτόν. Δεν θα μπορέσουμε να επεκταθούμε πολύ περισσότερο, μέχρι ότου θα έχει αποδειχθεί ότι πράγματι χρησιμοποιούνται αυτά τα στοιχεία και τα εργαλεία, ώστε να αξίζει η επένδυση πόρων σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Εξαρτάται λοιπόν από την χρηστικότητα και την αποτελεσματικότητα και θα δούμε στο μέλλον προσεχώς πώς αυτά μπορούν να επεκταθούν, να διευρυνθούν. Τώρα, γυναίκες και, οικονομίες, και οικονομία και τα συμπεράσματα. Τα όσα υπάρχουν και έχουν παραχθεί σε αυτό το πλαίσιο εξειδικευμένα, αυτό που κάνουμε είναι αναλύουμε με αυστηρό τρόπο επιστημονικά με βάση διάφορους δείκτες πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Αν είναι θετική η εξέλιξη θα υπάρχουν θετικά συμπεράσματα. Αν όμως οι δείκτες θα καταδεικνύουν μια αρνητική εξέλιξη πραγμάτων τότε τα συμπεράσματά μας θα είναι ε, φυσικά αρνητικά εντός εισαγωγικών θα αντανακλούν αυτή την πραγματικότητα. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα στατιστικά στοιχεία και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Αλλά επίσης ε, εκπονούμε ε, κύρια συμπεράσματα όπου προσπαθούμε να παρουσιάσουμε πιο φιλικά προς τους χρήστες, ε, με μια πιο φιλική προς τους χρήστες μορφή, πιο εύληπτη, που διευκολύνει τους χρήστες για όσους δεν έχουν και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να εξοικειωθούν και να αποκτήσουν μια ευρύτερη εικόνα. Λοιπόν, σίγουρα οπωσδήποτε θα έχουμε μέσα στα κυριότερα ουσιοδέστερα συμπεράσματα θα αναφέρουμε τα θετικά στοιχεία και εξελίξεις ε, και με τρόπο εύληπτο ώστε να ε, μην, ε, τα, μην αγνοηθούν. Αλλά και κάτι άλλο, στα κράτη-μέλη έχουμε συλλογή και εντοπισμό που προσπαθούμε να επιτύχουμε και σε σχέση με τα κράτη-μέλη για τις βέλτιστες προδιαγραφές. Και εδώ πάλι πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε αυτά με θετικό τρόπο βλέποντας πώς έχει επιτύχει ένα κράτος στο ένα ή το άλλο για την Ιταλική Προεδρία και μια εξειδικευμένη προσέγγιση ή και περιφερειακή προσέγγιση. Ενδιαφερόμαστε άμεσα για μια τέτοια περιφερειακή προσέγγιση με συμμετοχή των τοπικών αρχών, περιφερειακών αρχών. Θέλουμε να ε, μπορούμε να επικεντρωθούμε σε αυτό το επίπεδο πέρα από το ε, κεντρικό ε, επίπεδο Θέλουμε και οι τοπικές αρχές να μπορούν να, να συμμετάσχουν σε αυτή τη δυνατότητα σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία και τις συγκρίσεις τομεακά και επί των διαφορετικών θεμάτων. Έχουμε και επαφές και συζητήσεις και με την Eurostat, αλλά και με την Επιτροπή των Περιφερειών ως θεσμικό όργανο και με το ε, ε, όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τους Δήμους και τις Κοινότητες, ε, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Όλα αυτά σε ένα συγκρίσιμο πλαίσιο ευρύτερα που θα διασφαλίζει συγκρισιμότητα σε σχέση με τα κράτη-μέλη μεταξύ αυτών των στοιχείων και που με αυτόν τον τρόπο θα διατίθενται προς τα κράτη-μέλη. Απαιτεί περισσότερο χρόνο αυτό. Νομίζω η χρηματοδότηση που διασφαλίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από πρωτοβουλία που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εποπτεία αυτή τη ε, χάρτα ε, για την, ε, για την ισότητα των φύλων και σε σχέση και με τους δείκτες και άλλα στοιχεία έχουμε διαφορετικά κομβικά αλληλοσυνδεόμενα στοιχεία ως πρωτοβουλίες. Μόλις θα υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία και θα είναι διαθέσιμοι δείκτες και στοιχεία, με μεγάλη χαρά να τα, θα τα χρησιμοποιήσουμε. Και σε σχέση ε, με το gender-based violence, δηλαδή την βία σε σχέση με ε, το φύλλο, ε, ήταν δύσκολο να εξευρεθεί μια κοινή προσέγγιση. Πώς θα μπορούσε να μετρηθεί αυτή η πιο εξειδικευμένη σε σχέση με το κάθε φύλλο βία ε, πιστεύουμε ότι εφέτος θα τα καταφέρουμε και θα πετύχουμε να προχωρήσουμε. Η μέθοδος που υιοθετείται και χρησιμοποιείται είναι ότι θα προσπαθήσουμε να εκπονήσουμε κάποιους πρώτους δείκτες που θα αντανακλούν κάποια πράγματα. Είτε θα, δείχνει, θα δείχνουν τον ε, ισχυρό, την ισχυρότερη δεσπόζουσα παρουσία κάποιων ε, στοιχείων ε, όχι. Είναι δύσκολο να σας αναφέρω τα σχετικά γιατί δεν έχουν ε, ακόμα ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και να μπορέσουμε να αναλύσουμε για την εκστρατεία και ιδιαίτερα σε σχέση με το, το copyright, την διασφάλιση αυτού του, ε, το, πριν από 15 χρόνια από πλευράς κάποιου Καναδού ε, υπάρχει μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση σε σχέση με αυτή την πρωτοβουλία. Αν οι άνδρες δεν εξηγούν, δεν καθιστούν κατανοητό στους, άλλες, στους άλλους άνδρες ότι δεν μπορεί κανείς να δεχθεί ε, μια τέτοια κατάσταση, ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική υπόθεση, ότι είναι απαράδεκτη η βία κατά των γυναικών και ότι πρέπει κανείς ενεργά να εμπλακεί για να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο. Και νομίζω ο κύριος αυτός ήταν που ε, κατέβαλε αυτή την προσπάθεια υπέρ αυτών των ε, αξιών και πρωτοβουλίων και παγκόσμια. Σημαντικό είναι να συμμετάσχουμε κι εμείς σε αυτή την πρωτοβουλία. Διότι αυτό εξειδικεύει την πρωτοβουλία πώς άντρες μπορούν να πείσουν άλλους άντρες και ιδιαίτερα νέους να μην ασκούν βία και να μην εμπλέκονται σε τέτοια ε, συνάσκηση βίας κατά των γυναικών. Διαφορετικές δυνατότητες και μορφές δράσης πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Ε, αυτό είναι μόνο ένα μικρό τμήμα των δραστηριοτήτων μας. Ε, ίσως ε, μελλοντικά αυτή η εκστρατεία Gender Based Violence, GBV, η εξειδικευμένη προσπάθεια καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών θα μπορούσε να πάρει σάρκα και ωστά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ. Έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, Monsieur Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκφράζει την ικανοποίησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή τη σημερινή μας ε, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Ινστιτούτου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών του Κοινοβουλίου. Είναι καλό να υπάρχουν τακτικές επαφές, ακόμα πιο συστηματικές, μεταξύ του Ινστιτούτου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών, ώστε το Ινστιτούτο να κατανοήσει πλήρως το ρόλο που το αναλογεί ε, στα πλαίσια των ε, θεσμικών μηχανισμών και να καταλάβει καλύτερα τι στήριξη μπορεί να προσφέρει από τεχνικής πλευράς στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα εργασίας του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να σταθεί κυρίω στα όσα προβλέπονται να γίνουν για το θέμα τη βία κατά των γυναικών. Πρόκειται για έναν τομέα όπου πραγματικά το Ινστιτούτο μπορεί να προσφέρει προσθεθέμενη αξία. Να δημιουργήσει κάτι που δεν υπήρξε, ουδέποτε έγινε προηγουμένω στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Να τονίσουμε λοιπόν ξανά την ανάγκη να αναπτυχθούν ή να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη στατιστικών δεδομένων, ποσοτικών και για αυτό το θέμα. Ξέρετε ότι χωρίς μια συνοπτική θεώρηση, μια σφαιρική θεώρηση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι δύσκολο να κάνουμε μια συζήτηση που να βασίζεται σε συγκεκριμένε δεδομένα στην πράξη. Μια τεκμηριωμένη συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν το Ινστιτούτο καλά θα κάνει να συνεχίσει τις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, αναπτύσσοντας ή παροτρύνοντας να αναπτυχθούν στατιστικά δεδομένα και σε αυτό το θέμα. Η Επιτροπή βλέπει με ικανοποίηση ότι οι εκθέσεις για την Προεδρία του Συμβουλίου αυτή τη στιγμή έχουν περάσει στον ρυθμό της ρουτίνας θα έλεγα με δύο ετησίως εκθέσεις. Προς στιγμήν στο μέλλον θα προβλέπεται μία έκθεση ετησίως για να μπορέσει το Ινστιτούτο να έχει το χρόνο να ασχοληθεί και με άλλους τομείς. Οι εκθέσεις αυτές, και νομίζω ότι σωστά τονίστηκε σήμερα, Ιδίω η έκθεση για την ελληνική προεδρία περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Και ο δείκτης, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι μια πολύ σωστή πρωτοβουλία, ακόμη και αν θα πρέπει λιγάκι να συμπληρωθεί ή να αποσαφινιστεί. Πάντως πρόκειται για ένα εργαλείο που εδώ και κάπου, κάποιο καιρό α, περίμενε και ζητούσε να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή εδω και καποιο καιρο περιμενε και Γενικότερα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά καλεί τον Ινστιτούτο να συνεχίσει τις προσπάθειές του, πάνω απ' όλα για να συγκεντρώσει δεδομένα, δηλαδή να αναπτυχθεί η γνώση. Στη φάση αυτή όπου βρίσκεται το Ινστιτούτο μετά από τέσσερα χρόνια δραστηριοποίησης του, έκθεση, οι γνώσεις που συγκεντρώνουμε, τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα αποδεικνύεται ότι είναι εξαιρετικώς ε, χρήσιμα στο πολιτικό έργο του ε, Κοινοβουλίου και όχι μόνο του Συμβουλίου, και του Συμβουλίου μάλλον όχι μόνο σε επίπεδο Προεδριών, αλλά γενικότερα για το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έργο αυτό ε, είναι πολύ χρήσιμο στην πολιτική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή για την εκπόνηση της στρατηγικής το 2020 και σε ό,τι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την στρατηγική της ισότητας των γυναικών από την περίοδο για το 2010 έως το 2015. Ευχαριστώ. Okej, ε, tack så mycket för det. Och eh, då... Eh, eh. Ευχαριστώ για την ε, παρουσία σας και θα κλείσουμε εδώ τη συζήτηση για το σημείο αυτό. Ε, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που θα έχουμε συστηματικότερη συνεργασία, καλύτερα διαδρομένη και στο μέλλον. Και το έργο σας πραγματικά είναι καθοριστική σημασίας και για το δικό μας το έργο στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που ήρθατε σήμερα και ελπίζω ότι θα ξανάρθετε και θα μιλήσουμε πάλι για ενδιαφέροντα ζητήματα. Φυσικά και με ενδιαφέρει το θέμα αυτό, γιατί θα ήθελα να αποδειχθεί ωφέλιμη αυτή η συνεργασία και να έχω στα χέρια μου στο δυνατόν περισσότερο υλικό. Είναι λογικό αυτό για έναν πολιτικό. Πάντοτε αποζητούμε να έχουμε στο δυνατόν περισσότερου πόρου ε, ω προ την ενημέρωση και τι πληροφορίε. Αλλά είχαμε και πολύ χρήσιμη συζήτηση και διάλογο. Ε, και πραγματικά Εάν ε, η πραγματικότητα επέτρεπε να πούμε ότι έχουμε φτάσει στο 100% της ισότητας μεταξύ των φύλων, θα ήταν όλα πάρα πολύ ωραία, όμως αυτό δεν ισχύει ακόμη και γι' αυτό υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν. Και από τη δική σας πλευρά και από τη δική μας, αλλά και στη συνεργασία μας. Ευχαριστώ και πάλι λοιπόν για την προσέλευσή σας. Δεν ξέρω ακριβώς σε ποια ημερομηνία θα ξανάρθετε, αλλά θα είσαστε πάντοτε ευπρόσδεκτοι. Ευχαριστώ. Ωραία. Να προχωρήσουμε τώρα. Δεν ξεκινήσουμε αμέσως τις ψηφοφορίες, διότι στις 10 και 10 θα έρθει η κυρία Πακ και θα μας πει τι έγινε με την Επιτροπή Πολιτισμού, ε, γιατί μας επηρεάζει άμεσα η συζήτηση που έγινε εκεί να θυμίσω δύο πράγματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Όπως θα το γνωρίζετε, αύριο θα γίνει μια κοινή, μια μεικτή συνεδρίαση με την ε, Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στο ε, κτίριο Γιάν, στο 2Q2 για τις ειρηνευτικές Και βεβαίως είναι σημαντικό να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τα δικαιώματα των γυναικών σε καταστάσεις ένοπλων σειράξεων και τις εκθέσεις που έχει ετοιμάσει τις μελέτες που υπάρχουν σχετικά από τον ΟΗΕ. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ετοιμαστούν καλύτερα για το θέμα αυτό και θα είσαστε ευπρόσδεκτοι. Επίσης υπάρχει και άλλη μια εκδήλωση που προβλέπεται στις 5 Μαρτίου θεμελιώδη δικαιώματα και οργανισμός για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εκεί διοργανώνεται μία διάσκεψη όπου θα παρουσιαστεί μια έρευνα προς ενημέρωση του Συμβουλίου όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της, ε, των συνομιλιών και των συνεντεύξεων που υπήρξαν 41.000 γυναίκες. Μια έρευνα εξαιρετικής, εξαιρετικού ενδιαφέροντος για όλους τους συναδέλφους εδώ και πραγματικά θα μας ε, διευκολύνει πάρα πολύ και θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη για, για το έργο μας. Το απόγευμα λοιπόν της 5, της 5 Μαρτίου θα έχουμε και την ε, παρουσία Θα έχουμε την παρουσίαση ακριβώς αυτή του ΦΡΑ, του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, εν ώψη και της Παγκόσμιας ημέρας της Γυναίκας, 8 Μαρτίου. Σε αυτή τη φάση και επειδή θα πρέπει να καλύψω λίγο αυτό το χρονικό κενό, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία της παρουσίας της κυρίας Πακ. Θα μείνετε εκεί που είστε. Εφού, αφού φτάσατε, θα έχουμε και λίγο παραπάνω χρόνο. Οπότε σας δίνω πέντε λεπτά για την παρέμβασή σας και θα αρχίσουμε τις ψηφοφορίες στις 10 και 4. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Να σας πω κάτι ωραίο. Δηλαδή, όπως ξέρετε, υπάρχει το βραβείο Lux και συνήθως κέρδισε το μια ταινία που λέγεται ε, Η ξένη. Ε, και αφορά τα εγκλήματα τιμής. Ε, η, η ταινία αυτή έχει αναγνώριση, αλλά όχι επαρκή ακόμη και θέλουμε να την αξιοποιήσουμε για τον εξής λόγο. Στις 8 Μαρτίου ε, είναι η μέρα των γυναικών που θα είναι φέτος αφιερωμένη στη βία κατά των γυναικών. Και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και εγώ μαζί με την Άρτε, το κανάλι Άρτε, ε, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε. Ούτως ώστε θα παιχτεί στις 8 Μαρτίου η ταινία αυτή, στις 8 Μαρτίου λοιπόν, αλλά επί τρεις μήνες θα παίζεται επίσης στην διαδικτυακή πλατφόρμα ούτως ώστε όποιος θέλει να μπορεί για αυτούς τους τρεις μήνες να το κατεβάσει δωρεάν ε, σε όλες τις 24 γλώσσες της Ένωσης. Η ταινία αυτή, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα θαυμάσιο μέσο. Γι' αυτό έχω έρθει για να σας τα πω, ούτως ώστε οπουδήποτε είμεθα στις εκλογικές μας περιφέρειες ε, να μπορούμε να κάνουμε μια εκδήλωση με αυτή την ταινία είτε στην Εστονία, τη Γερμανία, στην Πορτογαλία, την Ελλάδα διότι θα υπάρχει δυνατότητα να κατεβάσει κανείς την ταινία σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες μας δωρεάν. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε έτσι ένα χειροπιαστό μέσο όλοι που δεν το είχαμε πριν. Είπα είναι δωρεάν. Και παρουσιάζει αυτό το θέμα των εγκλημάτων τιμής με έναν τρόπο που είναι πολύ συγκινητικός δεν προσπαθούμε λοιπόν να το κάνουμε με τρόπο ε, ιδιαίτερα επιθετικό, αλλά προσπαθούμε να δείξουμε τα διλήμματα αυτών που έχουν ε, ανατραφεί με αυτή την παράδοση και που ε, ακόμη και αν ζουν στο Βερολίνο σήμερα είναι υποχρεωμένοι, θεωρούν ότι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτή η ταινία έχει προβληθεί στην Τουρκία, στο Πακιστάν, εκεί που ζουν πολύ περισσότερο μουσουλμάνοι από ό,τι στις χώρες μας και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να αξιοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα. Είναι δωρεάν. Δωρεάν από την Άρτε στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Άρτε. Θα πάτε λοιπόν ε, στο arte.tv κάθετος Lux Minus Prize και σας διαβεβαιώ ότι θα, θα λάβετε όλη αυτή την πληροφόρηση και μέσω email γιατί βλέπω το δεν είναι πολλοί παρόντες. Ήθελα να έρθω λίγο πριν την ψηφοφορία για να με ακούσουν πολλοί συνάδελφοι. Αλλά είναι θαυμάσια λοιπόν η προσφορά. Σας παρακαλώ να την αξιοποιήσετε. Γιατί μας βοηθάει παντού στις εκλογικές μας περιφέρειες να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Έχουμε ευρωεκλογέ. Όλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική γυναικών και στη χώρα τους μπορούν λοιπόν να συγκινήσουν τους εκλογείς του. Νομίζω ότι είναι θαυμάσια πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πολύ την Άρτε που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Χαίρομαι πολύ που ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου υποστηρίζει αυτή την πρωτοβουλία και ελπίζω να αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία. Ξαναλέω, θα σας στείλω email για να τα έχετε όλα εύκολα και να μπορείτε να αξιοποιήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Πακ, σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε μαζί μας αυτές τις πληροφορίες. για ένα θέμα που μας αφορά άμεσα. Είναι πολύ εύστοχη η, παρα... η επισήμανσή σας και είναι και δωρεάν. Όχι μόνο εσείς βέβαια ως βουλευτές, οποιοδήποτε πολίτης έχει πρόσβαση όλες οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, ο Γιάννης, ο Γιώργος, όλοι μπορούν. Και μπορείτε και περαιτέρω να ενημερώσετε τις γυναικείς οργανώσεις, τις οργανώσεις βοήθειας προς τις γυναίκες. Νομίζω ότι θα τους βοηθήσει. Είναι μια δυνατότητα με την οποία μπορεί κανείς να μιλήσει και στους ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει με αυτή την παράδοση, να καταλάβουν το σφάλμα τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και πάλι, κύριε Πακ. Και από ό,τι κατάλαβα βεβαίως θα μας αποστείλετε την πληροφόρηση. Ωραία, πολύ ωραία. Ούτως ώστε και εμείς να μπορούμε να την ε, ε, διαδώσουμε περαιτέρω. Έχει κανείς ερωτήσει από αυτού. Όχι, ωραία. Ναι. Α, Είχα υποσχεθεί ότι 10 και 4 θα αρχίσουν οι ψηφοφορίε. Γιατί ξέρω ότι οι άλλοι είναι σε άλλε επιτροπέ. Λοιπόν, δεν θέλω να ενοχλήσω κανένα. Πέντε λεπτά διάλειμμα, αλλά παρακαλώ σε ακριβώς πέντε λεπτά να επανέλθετε. Τεσσερισήμιση λεπτά διάλειμμα. Τεσσεράμιση. Okay, uh, because I promised that we start vote 10:15. Λοιπόν, ε, θα αρχίσουμε την ψηφοφορία στις 10.15, έτσι υποσχέθηκα. Παρακαλώ καθίστε. Πρώτα το 4, οι διαπραγματεύσεις για τα, τις πολιτικές προοπτικες 2.14.20, διδάγματα και προοπτικές. Η συγγήτρια είναι η κυρία Ματέρα, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να παρευρεθεί. Νομίζω ότι θα την εκπροσωπήσει η κυρία Μπαστός. Οπότε σύντομα θα ε, μας ε, εξηγήσει η κυρία Μπάστος. If you want to take the floor. Εάν θέλετε να λάβετε το λόγο. Δεν θέλει. Εντάξει, τότε να προχωρήσουμε στις πληροφορίες Έχουμε πέντε τροπολογίες. Να τις ψηφίσουμε συνολικά, on block. Ωραία. Υπέρ, κατά, αποχές, να γκρίνονται. Περνάμε μετά στο 5 απαλλαγή του 2010 του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εδώ η κυρία Ματέρα είναι συγγήτρια αλλά η κυρία Μπαστός δεν θα πάρει πάλι το λόγο. Να ξεκινήσουμε με την τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. τροπολογία 2. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Με συγχωρείτε. Σωστά λέω τους αριθμούς, αλλά από λάθος κατάλογο. Να ξαναρχίσουμε. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά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 Να περάσουμε τώρα στο 6. Απαλλαγή 2012 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Ψηφίζουμε 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το ψήφισμα. Τελική ψηφοφορία άρχεται. Και πάλι το. Συγχαρητήρια στις συγκεκριές Σας ευχαριστούμε. Δεν υπάρχουν διάφορα. Δεν υπάρχει επιθέμα στα διάφορα. Οπότε θα συνεχίσουμε με τη συνεδρίαση των συντονιστών. Όμως οι συντονιστές θα συνεδριάσουν σε 5 λεπτά. Σε πέντε λεπτά θα αρχίσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα.